So, Αγαπητοί συνάδελφοι, καθίστε παρακαλώ. Ήδη μου είπανε ότι καθυστερώ και θα χάσω και τη φήμη μου. Wir Συζητήσεις δεν έχουμε σήμερα καθόλου. Διαπιστώνω ότι η μερίσια διάταξη εγκρίνεται λοιπόν όσο έχει προταθεί. Σήμερα έχουμε όλες τις γλώσσες στη διάθεσή μας εκτός από εστονικά, μαλτεζικά και σλοβακικά. Και από τις 9 μέχρι τις 12.30, αν χρειαστεί να πάει μέχρι τότε, υποδεχόμαστε και ε, μια ομάδα 20 τσέχων φοιτητών δημοσιογραφίας που θα παρακολουθήσουν όλη τη συνεδρίαση. Ο δεύτερος τριμερής διάλογος πρέπει να σας πω για την έκθεση Αντωνέσκου θα γίνει στο Στρασβούργο στις 4 Φεβρουαρίου, θα αρχίσει από εκεί. Και θα πάμε, αρχίζουμε. Σημείο 3 της ημερήσιας διάταξης, έκθεση Eckhout και το αποτέλεσμα του τριμέρους διαλόγου. Θα πρότεινα να κάνουμε μια δοκιμή. Βγάλτε παρακαλώ όλοι τις κάρτες ψηφοφορία σας για να ψηφίσουμε ηλεκτρονικά. Αρχίζει τώρα η ψηφοφορία για το αποτέλεσμα του τριμερούς διαλόγου. Κανονική ψηφοφορία. Ψηφίσατε όλοι. Ακόμα είναι ανοιχτή η ψηφοφορία. Πέρασε. So, 46. 46 υπέρ. Μερικοί απέχουν τρει και μία ψήφο κατά. Εγκρίνεται λοιπόν συγχαρητήρια και Eichhout. Συνεχίζουμε. Η επόμενη έκθεση τη κυρία Οκονή. Θα πρέπει να ψηφίσουμε για τη διαδικασία πρώτα. Θα πρότεινα να γίνει και αυτή ηλεκτρονικά. Αρχίζει τώρα η ηλεκτρονική ψηφοφορία. Τι ψηφίζουμε τώρα, τη διαδικασία πρώτα. Απόφαση επί της διαδικασίας γράφει. Τη διαδικασία ψηφίζουμε και μόνο πρώτα. Ψηφίσατε όλοι. Πέρασε. Εγκρίνεται λοιπόν. Και τώρα ηλεκτρονικά και πάλι. Unblock. Όλο μας λοιπόν το περιεχόμενο αρχίζει ηλεκτρονική ψηφοφορία και πάλι. Ψηφίσατε όλοι. und die abstimmung ist geschlossen. ist somit angenommen. Εγκρίνεται λοιπόν. Dann kommen Backloading und Ερχόμαστε στο backloading τώρα με αντιρρήσεις. Ψηφίζουμε την πρώτα η ένσταση ηλεκτρονικά. Αρχίζει η ψηφοφορία. Ψηφίσατε όλοι. Πέρασε. Απορρίπτεται. Για τη δεύτερη έσταση τώρα. Το δεύτερο ψήφισμα δηλαδή, θα ψηφίσουμε αυτή τη στιγμή, αυτή η ψηφοφορία. Ψηφίσατε όλοι. Abstimmung ist geschlossen. Πέρασε. Απερίφθηκε αυτό. Και τώρα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ζητάει να μειωθεί η περίοδος ελέγχου και πρέπει να το ψηφίσουμε. Το έχουμε συζητήσει με τους αδελφούς, Ψηφίζουμε τώρα λοιπόν. Ψηφίσατε όλοι. Πέρασε. Ist somit angenommen, beide Einsprüche sind abgelehnt. Απορρίπτονται λοιπόν και οι δύο αντιρρήσει ε, στάσεις και εγκρίθηκε ε, ε, το αίτημα για μείωση της περίοδου ελέγχου. Ωραία. Συνεχίζουμε. Στο σημείο 7 είμαστε της μέσης Δέταξης. Είναι η έκθεση του κυρίου Σκυλακάκη για τις εκπομπές διοξιδίου του άνθρακα από τις θαλάσσιες μεταφορές. Είστε έτοιμοι να αρχίσουμε. Πάμε. Ενοποιημένη πρώτη, consolidated ε, ηλεκτρονικά. Αρχίζει ψηφοφορία. Ψηφίσατε όλοι. Εγκρίνεται. Συνεχίζουμε. 117 τώρα είπε. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 115 B υπέρ κατά αποχές ηλεκτρονικά παρακαλώ ελέγχουμε την 115 B ψηφίσατε όλοι πέρα απερίφθη συνεχίζουμε ενοποιημένη τροπολογία 3 ηλεκτρονική ψηφοφορία κατευθείαν Αρχίζει. Ψηφίσατε όλοι. Πέρασε. Εγκρίνεται. 121 υπέρ. Κατά. Αποχές. απορρίψετε. 22 υπέρ. Dagegen. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Dann weiter bei mir mit vier. Στην 24 τώρα υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεν είναι σαφές. Ψηφίζουμε ηλεκτρονικά. Την 24 ελέγχουμε παρακαλώ. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας. Απορρίπτεται. 123 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Η ενωπημένη 2 ηλεκτρονικά αρχίζει ψηφοφορία. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας. Με μεγάλη πλειοψηφία εγκρίθηκε. 128 υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεν είναι σαφές. Ας ελέγξουμε παρακαλώ ότι είναι 128. Αρχίζει η ψηφοφορία. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας. Απορρίπτεται. 26. Φυσική του υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 27 και 129 είπε. κατά αποχές εγκρίνονται 28 είπε. κατά αποχές εγκρίνεται 130 και 323 είπε. κατά αποχές εγκρίνεται. Α, 131 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 29 υπέρ. Dagegen. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Ήτρε 12 Β, 132 Β. Μαζί και τις δύο υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 134 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίψεται. 135 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Ενωπημένη 4 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Και συνεχίζουμε τώρα στην 146, 147, 148, ή 14 και τραν 26, υπέρ όλου αυτού του μπλοκ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 149 υπέρ. Τσεκ. Ωραία ελέγχουμε όλες τις προηγούμενες 146 έως και 26 των μεταφορών ηλεκτρονικά άρχεται η ψηφοφορία. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας. Απορρίπτεται. 149 πέρα. Κατά. Απαχές. Απορρίπτεται. 150 και 327 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνονται. 32 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 33 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 151 και η 315 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 34, 152 και 16 ήτρα υπέρ κατά αποχές εγκρίνονται 153 και 37 17 κατά αποχές απορρίπτονται τραν 28 και 154 υπέρ κατά αποχές εγκρίνονται 35 υπέρ κατά αποχές εγκρίνονται 36 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 29 το μεταφορών σε τρία τμήματα. Τμήμα πρώτον υπέρ. Κατά. Αποχές. Τι είναι αυτή η δεξιά και πράσινη συμμαχία, έλεγχος αμέσως. Αρχίζει η ψηφοφορία για την 29 ηλεκτρονικά. Για την τραν 29 είπε. Ε, συγγνώμη, ψηφίσατε όλοι πέρας. Απορρίπτεται. 155 είπε. Όχι, όχι, έχουμε και δεύτερο τμήμα. Ζητάει συγγνώμη ο πρόεδρο. Συγγνώμη, το δεύτερο τμήμα τη 29 πρέπει να ψηφιστεί ακόμα είπε. Κατά. Αποχέ εγκρίνεται. 155 είπε. Κατά. Αποχέ εγκρίνεται. 37 είπε. Κατά αποχές εκρίνεται. 156 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 158 και 159 μαζί υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 30α υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 160, 161, 318 και 330 B. Κατά. Αποχές. Δεν είναι σαφές. Ψηφίζουμε όλο αυτό το σύνολο ηλεκτρονικά παρακαλώ. Αρχίζει τώρα η ηλεκτρονική υπολήθευση. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας. Εγκρίνεται. Δηλαδή απορρίπτεται διορθώνει ο πρόεδρος. 38 είπε. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 162 και 187 είπε. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 31 είπε. Κατά αποχές απορρίπτεται. 163 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. Τώρα συνεχίζουμε. Πάμε στη 41. Αλλάζουμε σελίδα. ψηφίπε. υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 158 τώρα. Υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 183 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται η 45 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται η 171 και οι υπόλοιπες καταπίπτουν διότι εγκρίθηκε η 45 και θα πάμε τώρα έτσι δεν είναι, ναι, εγκρίναμε τη 45, οπότε καταπίπτουν οι επόμενοι. Τώρα σας πω που θα πάμε. 192, σε μένα η σελίδα 12. 194 και 196, το βρήκαμε. 192, 194, 196, Κατά αποχές απορρίπτεται. Τώρα η 53 υπέρ κατά αποχές δεν είναι σαφές ας το ελέγξουμε ηλεκτρονικά παρακαλώ αρχίζει ψηφοφορή. ψήφισατε όλοι Abstimmung ist geschlossen. Okay. Mit dem Block ITRE e 30. Ήτρε 30α, 209, 210 και τραν 42 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 212 und Tran 212 και τραν 43 ε, υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Γενοποιημένοι 5 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται η 215, υπέρ κατά αποχές δεν είναι σαφές επαληθεύουμε λοιπόν τη 215 ηλεκτρονικά ψηφίσατε όλοι πέρας εγκρίνεται η 57 υπέρ κατά Αποχές εγκρίνεται. 44 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 45 σε δύο τμήματα. Τμήμα πρώτον υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Το δεύτερο τμήμα υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 2.16 και 3.31 είναι ταυτόσιμες υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 2.17 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 2.18 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 219 υπέρ κατά αποχές δεν είναι σαφές. Παρακαλώ να ελέγξουμε τη 219. Αρχίζει τώρα η ψηφοφορία. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας. Εγκρίνεται. Και συνεχίζουμε. 220 και 32 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Η 58. Όχι. Καταπέπτει αυτή. Έτσι δεν είναι. Όχι. Πρέπει να την ψηφίσουμε την 58. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 221. Τι θέλετε. Έλεγχο για την 58. Ηλεκτρονικά ψηφίσατε όλοι. Πέρας. Απορρίπτεται. 221 Υπέ κατά δεν είναι σαφές και αυτό θέλει η ηλεκτρονική επαλήθευση αρχίζει τώρα 221 ψηφίσατε όλοι πέρας εγκρίνεται 222 υπέ κατά αποχές απορρίπτεται 223 υπέρ. Κατά. Άποχες. Απορρίπτεται. 224 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Η τραν 46 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Τραν 47 σε δύο τμήματα. Τμήμα πρώτον υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται το δεύτερο τμήμα υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 225, 26, 27, ήτρε 33 και 348 όλο αυτό το πακέτο μαζί υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 228 υπέρ Dagegen. Κατά αποχές δεν είναι σαφές ηλεκτρονική επαλήθευση 228 αρχίζει τώρα Haben alle Ψηφίσατε όλοι πέρας. Δεν κρίθηκε. 229 υπέρ. Κατά. Μου δυσκολεύεται τη ζωή. 229 ηλεκτρονική επαλήθευση. Ψηφίσατε όλοι. Πέρασε. Εγκρίνεται. 230, Ήτρε. 230, Ήτρε 39 και 349 μαζί, είπε. Κατά. Αποχε. Δεν είναι σαφέστερη η ηλεκτρονική επαλήθευση αυτό. Αρχίζει τώρα η ψηφοφορία για τον μπλοκ αυτό. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας και απορρίπτεται ούτω. Συνεχίζουμε. Τραν 51 υπέρ. Κατά. Η Άννα Ρόσπαρ θα τιμηθεί, θα παρισμοφορηθει υπέρ, γιατί ήταν η μόνη που ψήφισε. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Τραν 53, αλλάζουμε σελίδα, υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Ήτρε 39. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 2.41. Και τραν 54. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 66. Όχι. Έχει καταπέσει. Μάλιστα. 2.42 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απερίφθη. Η συμβαστική 6 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Η τραν 56 υπέρ. Κατά. Άποχες δεν ψηφίζεται. Ηλεκτρονικά, συνεπώς, τραν 56 ηλεκτρονική επαλήθευση. Ψηφίζεται όλοι. Πέρασε. 55 <laughs> υπέρ και οι 55. Μα άμα δεν ψηφίζετε, ε, Ρίχαρτ Ζέμπερ, σηκώστε κανένα χεράκι. 245 υπέρ. Όχι, όχι, έχει καταπέσει, λάθος. Συγγνώμη, πρόεδρος. Τραν 57, υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Τραν 58, υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Ήτρε 42 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 69 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Οι 250 ή 343 καθώς και τραν 59 μαζί. Και οι 111. Υπέρ. Κατά. Αποχές δεν είναι σαφής αυτό. Όλο αυτό το μπλοκ ηλεκτρονικά θα παληθεύουμε. Τώρα ψηφίσατε όλοι. Πέρασε. Απορρίπτεται. 19 των μεταφορών. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 253 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Λιτράν 60 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 254 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 255 πε κατά αποχές απορρίπτεται 256 πέ. κατά αποχές απορρίπτεται 257 είπε, κατά αποχές εγκρίνεται 70 είπε, κατά αποχές εγκρίνεται 259 επέ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται 260 επέ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται 261 επέ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Ή 262 επέ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται 263 επέ. Καλά. Κατά εποχές απορρίπτεται 264 υπέρ κατά εποχές απορρίπτεται 265 υπέρ κατά εποχές 266 υπέρ κατά εποχές απορρίπτεται 71 υπέρ κατά εποχές εγκρίνεται 267 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 268 υπέρ κατά αποχές δεν είναι σαφές και χρειαστεί ηλεκτρονική επαλήθευση αρχίζει τώρα για 268 ψηφίσατε όλοι πέρας Ist abgelehnt. Απορρίπτεται. 72 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 269 και όχι. Καταπίπτει. 271 υπέρ. Dagegen. Κατά. Αποχές. Απορρίφθηκε. 73 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 272 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Ήτρε 1. Είναι στη σελίδα 23 στο κατάλογο μου υπέρ. Ήτρε κατά αποχές απορρίπτεται 2 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται ήτρε 2 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται η 3 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 4 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται τραν 1 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται Τραν 2 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Η 6 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Η 4 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Η 7 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τραν 3 πίπτη Πάμε στο συμβεβασμό 7 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται η 9 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 83 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται τραν 6 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 85 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται η 7 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Η 8 υπέρ. 8. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 86 υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεν έχω καταλάβει. Ας την έλεξουμε ηλεκτρονικά. 86 αρχίζει ψηφοφορία. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας. Εγκρίθηκε. Και τώρα συνεχίζουμε. Τραν 12 γυρίζουμε σελίδα υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Η 16 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 100 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 17 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 102 και 314 μαζί Είπε. κατά αποχές δεν είναι σαφές ελέγχουμε την 102 και 314 ηλεκτρονικά αρχική ψηφοφορία ψηφίσατε όλοι πέρας απορρίπτεται 101 είπε. κατά αποχές απορρίπτεται 103 επέ κατά εποχές εγκρίνεται 104 επέ κατά αποχές απορρίπτεται 36 υπέρ κατά Αποχές απορρίπτεται. Ήτρε 6, ήτρε 7 μαζί. Υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Η 84 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 106 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 105 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Η τρενέα υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Η 108 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Η 109 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται 19 ο υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται τώρα πάμε στις τελικές ψηφοφορίες πάντα ηλεκτρονικά πρώτα θα ψηφίσουμε την πρόταση όπως τροποποιήθηκε αρχής ψηφοφορία. ψηφίσατε όλοι Πέρασα. 41 υπέρ, 9 κατά, 7 αποχές εγκρίθηκε. Τώρα, το νομοθετικό ψήφισμα θα ψηφίσουμε, αρχή υποφορία. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας. Εγκρίθηκε 44 υπέρ, 6 ε, κατά και 5 εποχές. Συγχαρητήρια κύριε Σκυλακάκη. Θέλετε να αρχίσουμε τις διαπραγματεύσεις για ε, συμφωνία σε πρώτη ανάγνωση. Ναι, θα ήθελα να ζητήσω εντολή ώστε να μπορέσουμε να καταφέρουμε να καταλήξουμε σε κάποιο αποτέλεσμα πριν τελειώσει η θητεία. Χρειαζόμαστε 36 ψήφους, γι' αυτό και ψηφίζουμε ηλεκτρονικά, αρχίζει τώρα η ψηφοφορία. Ψήφισατε όλοι. Δύο συνάδελφοι ακόμα να ψηφίσουν παρακαλώ. Πέρας. 44 είπε 10 κατά. Χωρίς αποχές. Ωραία. Θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους τους όλους Ευχαριστώ. Και εγώ εσάς ε, και συγχαρητήρια κύριε Σκυλακάκη. So. Ο Κρήτον Ασθένης έχει το λόγο. Procedural issue. Ένα διαδικαστικό θέμα. Πολύ σημαντική η απόφαση που ελήφθη σήμερα και συγχαίρω τον κύριο Συγγετή εκ μέρου των σοσιαλιστών. Αλλά τώρα έχουμε την ελληνική προεδρία που πρέπει να κάνει όλη τη δουλειά και να επιταχύνει τη διαδικασία. Ξέρουμε ότι είναι ένα πολύ σημαντικό θέμα για την Ελλάδα και ελπίζω ότι αυτό θα αποτελέσει κίνητρο για να εργαστούμε πιο σκληρά και πιο γρήγορα. Ευχαριστώ. Πιο σκληρά, πιο γρήγορα, μάλιστα. Αλλάζουμε τώρα θέμα. Πάμε στον Πίτερ Λίζε. Και αρχίζουμε την ψηφοφορία για την έκθεση Λίζε. Καταρχάς ψηφίζουμε ηλεκτρονικά για την συμβαστική πρόταση 1. Πίτερ Λίζε, έχεις τον λόγο. Ναι, ε, αν δεν κάνω λάθο, ο Μπά ότι έχει υποβάλει μια αίτηση απόρριψη όλη τη έκθεση, την οποία απορρίπτω και αυτό δεν καλούμαστε να ψηφίσουμε. Και μου λείπει το πλήν για αυτή την ε, συμβαστική τροπολογία και το συμφισικά και τη δική μου. Ναι, λέει ο πρόεδρο, εγώ έχω δει μόνο αυτό εδώ το κίτρινο κουτί και εκεί κοίταξα. Έχει φυσικά δίκαιο ο εισηγητή. Ψηφίζουμε καταρχά για την ε, τροπολογία 21. Υπέρ, κατά αποχές απορρίπτεται λοιπόν. Περνάμε τώρα στην συμβαστική τροπολογία 1. Ηλεκτρονικά παρακαλώ, άρχεται η ψηφοφορία. Ψηφίσατε. Πέρας. 33 ψήφοι υπέρ, 15 κατά, 7 αποχές. Προχωράμε. Συμβιβαστική 2. Επίσης ηλεκτρονικά άρχεται η ψηφοφορία. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας. 41 ψήφοι υπέρ, 13 κατά εγκρίνεται λοιπόν. Συνεχίζουμε με την 74 υπέρ. Στη σελίδα 5 όπως το βλέπω. Υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. ενοποιημένη 3 υπέρ. Ή ηλεκτρονικά θα το κάνουμε, συμβαστική 3. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας. Στη σελίδα 10. Πέρας. Εγκρίνατε. Περνάμε λοιπόν στην συμβαστική 4. Επίσης ηλεκτρονικά άρχεται η ψηφοφορία. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας. Εγκρίνεται. Αιτιολογικές σκέψεις τώρα. 22. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 1. Ήτρε. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Χόλγκερ Κράμερ. 23. Υπέρ κατά, αποχές, απορρίπτεται. Τραν 1, υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 2, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 25 και 2 μαζί, υπέρ. Κατά, αποχές, απορρίπτονται. 27. Κράμερ. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 26. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Συμβιβαστική 6. Η ηλεκτρονικά άρχεται η ψηφοφορία. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας. 52 ψήφοι υπέρ, 4 κατά. 1 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 29. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Πάμε τώρα στην 30, 31, 32 και 3. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτονται. 4. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 34. Υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 3. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 35. Υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 33. Υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Όχι, καταπίπτει. Δεν χρειάστηκε να την ψηφίσουμε λοιπόν. 5. Συμβαστική 5. Ηλεκτρονική ψηφοφορία άρχεται. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας εγκρίνεται. 42 ψήφοι υπέρ, 13 κατά. 7 υπέρ, κατά. Αποχές εγκρίνεται. 36 και 37 και 38, 8 και 4. Όλες αυτές μαζί υπέρ, κατά. Αποχές απορρίπτονται. 39 τώρα, 40... Δεν ακούγεται η μετάφραση προς τα πολωνικά. Δεν ακούγεται η πολωνική διερμηνία. Τώρα, ναι, τώρα ακούγεται. 39 λοιπόν, 40, 41, 42 και η 35. Υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτονται. 44, 45, 46, 9 και 6 υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτονται. 5 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 47, 10 και ήτρε 7 υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. 6 υπέρ, κατά, Αποχές εγκρίνεται. 49. Υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Περνάμε λοιπόν στην πρώτη τελική ηλεκτρονική ψηφοφορία. Άρχεται. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας. Εγκρίνεται με 40 ψήφους υπέρ, 8 κατά και 6 αποχές. Δεύτερη ψηφοφορία, τελική, ηλεκτρονικά για το νομοθετικό ψήφισμα. Είπε, άρχεται η ψηφοφορία. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας. Επίσης εγκρίνεται. Και τελειώνουμε την ψηφοφορία. Ο εισηγητή θα ήθελε διαπραγματευτική εντολή. Ο Κρι Εύης όμως έχει ζητήσει το λόγο. Παρακαλώ. Κύριε Πρόεδρε, Γνωρίζουμε ότι η διαδικασία Stop the Clock επιβάλλει χρονικά όρια, οπότε υποστηρίζουμε το να δοθεί θητεία στον εισηγητή, αλλά αυτό ανατρέπει τη γνωμοδότηση δύο άλλων επιτροπών και θεωρώ ότι αν οι κανόνες του Κοινοβουλίου λειτουργούσαν κανονικά, το Κοινοβούλιο θα έπρεπε να μπορεί να έχει μια ευκαιρία να κάνει μια απόφαση συνολικά. Δεν έχω πρόβλημα να υποστηρίξουμε, αλλά θεωρώ ότι η διαδικασία είναι μη δημοκρατική. And the rules of procedure should be changed. Και θα πρέπει να αλλάξει ο εσωτερικός κανονισμός. Να απευθυνθείτε στον συνάδελφο Νταφ. Όμως δυστυχώς δεν μπορούμε να το συζητήσουμε αυτό εδώ. Ο εισηγητής έχει το λόγο. Ευχαριστώ πολύ πρόεδρε. Πράγματι βρισκόμαστε σε μια δύσκολη θέση δεν μπορούμε να πάμε στην Ολομέλεια, διότι υπάρχει ο κίνδυνος να μην καταφέρουμε να αλλάξουμε την νομοθεσία και να μην είμαστε ευχαριστημένοι με το αποτέλεσμα. Πάντως πιστεύω ότι δεν θέλουμε να επανέλθει η αρχική νομοθεσία για τις ε, υπερατλαντικές πτήσεις. Έχουμε συμπεριλάβει στοιχεία και προτάσεις από την Επιτροπή Μεταφορών Η Τραν, λοιπόν, θα είναι παρούσα στον τριμερή διάλογο. Δεν μπορούμε τώρα να αλλάξουμε τα πράγματα, όπως σας είπα. Ε, μπορώ να στηρίξω... Ζητώ όμως να στηρίξω τη διαπραγματευτική εντολή, διότι διαφορετικά δεν θα προλάβουμε να ολοκληρώσουμε το νομοθετικό μας έργο μέχρι τον Απρίλιο. Ο Μπάς Αίκαουτ πρότεινε να απορριφθεί στο σύνολό της η πρόταση αυτό όμως το καταψήφισε η Επιτροπή, διότι δεν ήμασταν όλοι 100% σύμφωνοι για το πώς θα βρούμε ένα συμβιβασμό. Ζητώ όμως να με στηρίξετε, διότι είναι καλύτερο αυτό και προτιμότερο από το να απορρίψουμε γενικά την πρόταση. Μάλιστα λοιπόν, ο εισηγητής ζητά διαπραγματευτική εντολή και την ψηφίζουμε. Άρχεται η ψηφοφορία. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας. 49 ψήφοι υπέρ, 6 κατά, μία αποχή. Πίτερ Λίζε, Σας εύχομαι ως εισηγητής να έχετε επιτυχία. Τη χρειάζεστε. Ευχαριστώ και τους συναδέλφους για την πολύ συγκεντρωμένη δουλειά τους. Προχωράμε τώρα με το σημείο 9. Παύλ Ποκ, Έχετε όλοι τους καταλόγους μπροστά σας για την ψηφοφορία. Ναι, μπορούμε να αρχίσουμε. 106 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 107-108 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτονται. 109 υπέρ. Κατά. Αποχές δεν είναι σαφές. Ηλεκτρονική επαλήθευση για την 109. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας. Εγκρίνατε. 110. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνατε. Είχα 111 κατά πίπτη. Περνάμε στην ενοποιημένη 5. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνατε. τα 9. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 113. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 115. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 114. Κατά τμήματα. Πρώτο τμήμα. Υπέρ. Κατά. Άποχες. Απορρίπτεται. Δεύτερο τμήμα. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεν είναι σαφές. Η ηλεκτρονική επαλήθευση για το δεύτερο τμήμα της 114. Άρχεται η ψηφοφορία. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας. Οι σοσιαλδημοκράτες έχουν μία ψήφο παραπάνω. Επαναλαμβάνουμε. Δεύτερο τμήμα λοιπόν της 114. Ηλεκτρονική επαλήθευση. Άρχεται η ψηφοφορία. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας. Απορρίπτεται. Εκατόν δεκαπέντε. Υπέρ. Κατά. Αποχές. 15. Ηλεκτρονική επαλήθευση. Άρχεται η ψηφοφορία. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας. Απορρίπτεται. Είναι τα 10. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνατε. 116. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 117. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 118. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Έχουμε νέο συνάδελφο στην πρώτη σειρά.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 Συμβιβαστική 1. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 139. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεν είναι σαφές. Η ηλεκτρονική επαλήθευση για την 139. Άρχεται η ψηφοφορία. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας. Απορρίπτεται. 140. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Πες 7 υπέρ. Κατά. Άποχες απορρίπτεται. 17 και 19 μαζί υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνονται. Δεκαοχτώ υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 142 υπέρ. Κατά. Αποχές δεν είναι σαφές. Η ηλεκτρονική επαλήθευση για την 142. Άρχεται η ψηφοφορία. Ψηφίσατε όλοι. Πέρασε. Εγκρίνεται. Είναι τα 13. Υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 144 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Είναι τα 14 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 146 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Περνάμε τώρα Στην ΠΕΣ 9. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 147. Υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 148. Υπέρ. Κατά. Αποχές δεν είναι σαφές. 148 ηλεκτρονική επαλήθευση. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας. Απορρίπτεται. 149 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 150 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 151 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 21 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 153. Υπέρ. Κατά. Άποχες απορρίπτεται. 154. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 155, 156, 157, ίντα 17, πες 11. Όλες αυτές μαζί υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνονται. 160 υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. Ενοποιημένοι 2 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική 8 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 22 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 3 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 28 στη σελίδα 7 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Ενοποιημένη 4 υπέρ Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 218-223 στη σελίδα 9, όπως τη βλέπω, υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτονται. 219, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 220-225 υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτονται. 221 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 224 υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. Ηλεκτρονική επαλήθευση για τη 224. Έχει στηθεί, άρχεται η ψηφοφορία. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας. Απορρίπτεται. 234. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 40. Υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. 237 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 238 υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. 239 υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. 240 υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. 41 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 2.41, 2.44, 2.47, 2.49. Υπέρ. Κατά. Αποχές δεν είναι σαφές η ηλεκτρονική επαλήθευση. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας. Εγκρίνονται. Προχωράμε στην 246. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Ξανά άλλη μια φορά. 2.46. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 2.48. Υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 250 καταπίπτει. 2.52. Υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. 42 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 253 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 254 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 255 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 43 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Ίντα 20 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 257. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 258. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 259. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 260. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 261. Υπέρ. Κατά. Αποχές Απορρίπτεται. 262. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 264. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. τα 21. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 265. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 267. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 268. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 269. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 270. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 271, 72, 71 και 72 είναι ταυτόσιμες υπέρ, κατά, απορρίπτονται. 2,73 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 2.74 υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. 44 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 2.78 υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. 2.79 υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. Είναι τα 23 υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. 2.80 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 2.81 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 2.82 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 2.83 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Ενοποιημένη 7 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 291 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 293 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Πες 17 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 294 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. τα 24 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 295 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. Πες 18 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 2.96 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 2.97 υπέρ η ηλεκτρονική επαλήθευση για την 296. Άρχεται η ψηφοφορία. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας. Εγκρίνεται. Πάλι καλά που το κοιτάξαμε. 47, 48, 49, 50, 51, όλες μαζί. Υπέρ, κατά, εγκρίνονται. 2,98. Υπέρ, κατά, απορρίπτεται. 52. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Στην 306 περνάμε. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Ενοποιημένη 9. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 56. Υπέρ. Κατά. Εγκρίνονται. 318. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 319. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 320. Υπέρ κατά, αποχές, εγκρίνεται. 324 υπέρ, κατά, εγκρίνεται. 326 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 327 υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται 328, Κατά καταπίπτει 328 και 329. Αιτιολογικές σκέψεις 57 υπέρ, κατά, αποχές, δεν είναι σαφές, ηλεκτρονική επαλήθευση για την 57. Άρχεται η ψηφοφορία. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας. Εγκρίνεται. Ένα. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 58 και 59 υπέρ. Κατά. Εγκρίνονται. 60 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 61 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 62 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 63 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Είναι τα 1 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 64. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Περνάμε στην 68, επόμενη σελίδα. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 3. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Είναι τα 3. Υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 69 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Πες 2 υπέρ κατά αποχές εγ... απορρίπτεται. 71 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 72 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 73 υπέρ κατά Απορρίπτεται. Τι είναι αυτό, συναγερμός, πιάσαμε φωτιά, Twitter. Τέσσερα. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Πες τρία. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Είναι τα πέντε. Υπέρ κατά, αποχές, δεν είναι σαφές. Ξανά, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 78, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Πες 4, υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 105, υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Είναι Υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 5. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Και είναι τα 6. Επίσης πάμε στην 80. Υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 6. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 81. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 82. Υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. τα 7. Υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 83. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 84. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 7. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 86. Υπέρ κατά, αποχές απορρίπτεται. 88 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 91 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 92 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 9 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 93 υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. 10 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 94 υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. 94 ζητήθηκε ηλεκτρονική επαλήθευση. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας. Εγκρίνεται. Συγχαρητήρια. 96 96. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 97. Ε, υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 98. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 101. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 102 υπέρ, κατά, εγκρίνεται. Καταπίπτουν οι επόμενε. Περνάμε στην πρώτη τελική ηλεκτρονική ψηφοφορία. Άρχεται η ψηφοφορία. Ψηφίσατε. Πέρας. 50 ναι, 1 όχι, 5 αποχές. Περνάμε έτσι λοιπόν στην δεύτερη τελική ψηφοφορία. Άρχεται η ψηφοφορία. Ψηφίσατε. Πέρας. 49 ναι, 4 όχι, 3 αποχές. Και ρωτώ λοιπόν τον εισηγητή, θα θέλατε εντολή. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να ζητήσω από την Επιτροπή εντολή για να ξεκινήσω το με του Συμβουλίου και θα ήθελα να ευχαριστήσω και όλους τους συνεισηγητές. Η συνεργασία μας ήταν πολύ καλή και σοβαρή. Ευχαριστώ. Ωραία. Λοιπόν, ψηφίζουμε για την ανάθεση διαπραγματευτικής εντολής. Χρειαζόμαστε 36 θετικές ψήφους. Άρχεται η ψηφοφορία ηλεκτρονικά. Ψηφίσατε. 46 θετικές, 7 αρνητικές. Συγχαρητήρια λοιπόν, Παύελ Ποκ. Μπράβο σας, καλή τύχη. So, jetzt geht's weiter. Συνεχίζουμε. Είμαστε στο σημείο 10 τη ημερησία διάταξη. 3 και 4 μαζί οι τροπολογίε. υπέρ, κατά. Εποχές εγκρίνονται. 2 μέχρι και 10 υπέρ, κατά. απόχέ εγκρίνεται. Αμπλοκ πάλι. 11 με 13 υπέρ, κατά. Αποχές εγκρίνονται. Η 1 υπέρ, κατά. αποχέ εγκρίνεται. Πρώτη ηλεκτρονική ψηφοφορία, η πρόταση όπως τροποποιήθηκε, αρχίζει τώρα. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας. Εγκρίνεται. Δεύτερη ηλεκτρονική, αρχίζει η ψηφοφορία. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας. Κάτι έχω ακούσει ότι ο εισηγητή θέλει να αρχίσει διαπραγματεύσεις με το Συμβούλιο και θα πρέπει να ψηφίσουμε για να του δώσουμε την εντολή. Αρχίζει τώρα η ψηφοφορία. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας. Μάλιστα. Ευχαριστώ πολύ όλους ε, τους παρόντες και όλους όσοι συνεργάστηκαν σε αυτό το θέμα για την επικοδομητική μας συνεργασία. Και συνεχίζουμε. Στο σημείο 11 είμαστε τώρα. Ψηφίζουμε τη γνωμοδότηση της κυρίας Αντωνέσκου. Έχουμε την τροπολογία 4. Ψήφι υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 33 υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεν είναι σαφές. Χρειάζεται ηλεκτρονικό έλεγχο. Αρχίζει τώρα η ψηφοφορία. Haben abgestimmt? Ψηφίσατε όλοι. Πέρας. Απορρίπτεται. Dafür. Πέντε υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 34 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 35 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 36 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 37 είπε, Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 38 είπε, Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Η 6 είπε, Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Η 7 είπε, Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 39 είπε, Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 8 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 40 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 41 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 42 υπέρ κατά αποχές ε, απορρίπτεται 9 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται η 10 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 43 επε κατά αποχές. Τι ήταν αυτό τώρα. Μπορεί να μην πει κάποιο τι ψηφίσαμε. Ας το ελέγξουμε καλύτερα. Αρχίζει για τη 43 ηλεκτρονική επαλήθευση. Εγώ δεν είδα τι έγινε. Πέρας. Α, σαφέστατα εγκρίθηκε μαζί τις επόμενες 44 και 49 υπέρ. Κατά. Άποχες εγκρίνεται. Η 11 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Η 45 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 12 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Η 48 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 50 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται η 51 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 52 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 53 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται η 54 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται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 ή 19 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 20 κατά πίπτη 21 υπέρ 19 την εγκρίναμε μάλιστα έχετε δίκιο 20 πρέπει να ψηφιστεί ψηφίζουμε την 20 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 21 κατά αποχές εγκρίνεται 22 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 23 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 24 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 25 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 26 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 27 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 28 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται η 1 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται η 2 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 29 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται η 30 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται η 3 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 31 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 32 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται ηλεκτρονική τελική ψηφοφορία. Άρχεται, ψηφίσατε όλοι. Πέρασα. 50 υπέρ, κανείς κατά μία αποχή, συγχαρητήρια στην εισηγήτρια. Συνεχίζουμε. Έχουμε το σημείο 12 τώρα. Είναι η γνωμοδότηση του κυρίου Σόνικ Η 16 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. Η 3 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 17 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 18-19 μαζί υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. Η 4 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται είπε 5, 6, 7 μαζί είπε ορίστε τι θα ψηφίσουμε τώρα όμως Α, sie sind, sie sind Α, είναι συμβατές. Μπορούμε να τις ψηφίσουμε μαζί ή ξεχωριστά. Ξεχωριστά. 5 είπε. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Η 6 είπε κατά αποχές εγκρίνεται 7 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται η 1 καταπίπτει 8 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 9 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 10 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται η 11 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 2 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 12 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 13 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 14 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 15 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται τώρα πάμε στην ηλεκτρονική τελική αρχίζει η ψηφοφορία ψηφίσατε όλοι παρακαλώ Πέρας. είπαμε. 47 υπέρ, κανείς κατά τρεις αποχές, συγχαρητήρια κύριε Σόνικ. Και ερχόμαστε στην επόμενη ψηφοφορία, είναι το σημείο 13 στην ημερησία διαταξή. 49 σελίδες δεν είναι τίποτα ο κατάλογος ψηφοφορίας. Ε, μπορούμε να το κάνουμε και πιο σύντομα. 75, 76, 78 και 80 μαζί μπορούμε να τις ψηφίσουμε ηλεκτρονικά. Αρχίζει η ψηφοφορία. Ηλεκτρονικά. Haben Ψηφίσατε όλοι. Ένας ακόμα. Πέρας. 46 υπέρ, 4 κατά. Οπότε το διεκπαιρεώσαμε, το έχουμε επαναπέμψει και ε, ψηφίζουμε, ε, την τελική τώρα ψηφοφορία έχουμε για τη γνωμοδότηση. Παρακαλώ και εδώ ηλεκτρονικά. Αρχίζει η ψηφοφορία. Ψηφίσατε όλοι. Ψηφίσατε όλοι. Πέρα. Έληξε. 49 υπέρ, χωρίς αποχές. Είναι σαφέστατο. Εκφράσαμε με όσο μεγαλύτερη σφοδρότητα γινόταν τη δυσφορία της Επιτροπής μας. Ε, αυτά. Δεν έχουμε τίποτα άλλο πια στην ημερήσια διάταξη. Επόμενη συνεδρίαση στις 12 Φεβρουαρίου 9 με 12.30 και 3 με 6.30. Στις 13 Φεβρουαρίου 9 με 12.30 και 3 με 6.30 το απόγευμα. Ε, συνήθισε εδώ της Επιτροπής. Πέτερ Λίζε. Να κάνουμε τώρα μέσω συντονιστές. Παρακαλώ όσοι δεν είστε συντονιστές να αποχωρήσετε και οι υπόλοιποι να παραμείνουν για να διεκπαιρεώσουμε αμέσως και τη συνεδρίαση των συντονιστών.